σημείο της σημερινής διάταξης είναι σύντομη εισήγηση εκθέσεως Harbor. Προεμπορικέ δημόσιε συμβάσει, πρόθεση και καινοτομία στην εξασφάλιση βιώσιμων και ποιοτικών δημοσίων υπηρεσιών στην Ευρώπη. Έχει το λόγο, κύριε Χάρμπορ. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευτυχώ που έχουμε εδώ την κυρία Ρέντινγκ από την Κομισιόν απόψε, διότι η έκθεσή μου ασχολείται με μια πρόταση που εξελίχθηκε σε συνεργασία και διαμορφώθηκε με τις δικές της υπηρεσίες τόσα χρόνια. Πάρα πολύ σημαντική υπόθεση και έχει επίσης μακρόπνοες συνέπειες για το σύνολο της Ένωσης και της οικονομίας της Ευρώπης. Πρώτα πρώτα όμως να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες της κυρίας ε, ε, Ρέντιν. Θα πρέπει όμως θα πρέπει να ασχοληθούν ευρύτερα με το θέμα, να διαδοθεί η προβληματική αυτή, μια που περνάμε τέτοιου δύσκολου οικονομικού καιρού. Ποιο είναι το θέμα, ποιο είναι ο πυρήνα του ζητήματο, είναι πρόεδρε, ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι αρχέ δαπανούν για προϊόντα και υπηρεσίες πάρα πολλά χρήματα. Ένα 800 δις δαπανάτε για αυτές τις δημόσιες συμβάσεις και πόσα τελικά πηγαίνουν όσον αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη για νέες λύσεις για όλες αυτές τις προκλήσεις και όλα αυτά που αντιμετωπίζουν οι αρχές κάθε μέρα. Καλύτερες υπηρεσίες υγείας, καλύτερες υπηρεσίες ε, μεταφοράς, αλλαγή κλίματος, ενεργειακά αποτελεσματικά κτίρια. Λιγότερο από το 1% είναι η αναλογία αυτών των χρημάτων για τι δημόσιε συμβάσει για αυτά τα ζητήματα. Άρα, σα παραπέμπω στην συνθήκη τη Λισαβόνα και στο στόχο του 3%. Πάρα πολλέ δυνατότητε εκμετάλλευτε υπάρχουν εδώ ακριβώ σε αυτό το σημείο. Αναδύεται η έννοια τη προεμπορική δημόσια σύμβαση. Με ευθύ τρόπο θα πρέπει να γίνεται έρευνα να να τονώνουν την ζήτηση για τέτοιες λύσεις κυρίως από τις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις γιατί αυτοί κυρίως θα ωφεληθούν από τέτοιες προεμπορικές δημοσιοβάσεις. Μπορούν να προβλέψουν και εκεί που δεν υπάρχουν ακόμα εμπορικές λύσεις να τις αναζητούν, να τις δημιουργούν. Όμως θα πρέπει η έρευνα για ανάπτυξη σε αυτό τον τομέα να χρηματοδοτείται από το δημόσιο. Και αυτές οι λύσεις να πηγαίνουν στην επόμενη φάση που θα είναι οι βιώσιμες τέτοιες υπηρεσίες και προϊόντα. Ήδη έχουμε κάποια εμπειρία για κάποιες επιχειρήσεις που έχουν χρησιμοποιήσει τέτοιου είδους πόρους και έτσι μπόρεσαν να διαμορφώσουν κάποια αποδοτικά προϊόντα. Lead Market λέγεται αυτή η πρωτοβουλία της κυρίας, της κυρίας αγοράς και αφορά μεταφορές, αλλαγή κλίματος, υγεία. Και μέσω της εκθεσής μου ζητώ να υπάρχει περισσότερη κατάρτιση, να βάλουμε περισσότερο υπόψη την άριστη πρακτική και άρα αυτές οι προτάσεις να γνωρίσουν μεγαλύτερη διάδοση. Παρακαλώ και εύχομαι το κολέγιο των επιτρόπων αυτό να το λάβει υπόψη και ενεργήσει ένα λόγος και εν κατακλεί θα πρέπει να σας πω και επιτρέψτε λίγο παραπάνω χρόνο πρόεδρε για να τονίσω να τονίσω σε αυτή την άδεια ότι ήδη έχουμε δύο εκθέσεις από την Νομική Επιτροπή και από την Βιομηχανική Επιτροπή που δεν μπορούμε τώρα εδώ να τις ε, παρουσιάσουμε γιατί θα βοηθούσαν. Ευχαριστώ όμως ε, τον κύριο Χάση τον σκιώδη συγητή για τη δουλειά του. Οπότε Εν κατακλείδη θα σας πω ότι όλοι θα βγουν κερδισμένοι από αυτή την πρόταση και η κοινωνία και οι πολίτες και το δημόσιο και οι επιχειρήσεις και όσοι ασχολούνται με την γενοτομία και κυρίως η ευρωπαϊκή οικονομία και γι' αυτό και αυτή η υπόθεση είναι τόσο σημαντική. Και θέλουμε να συνεχίσουν τις επενδύσεις τους οι δημόσιες αρχές παρά τους δύσκολους καιρούς οπότε αυτή η πρόταση τώρα έγινε ακόμα πιο σημαντική από όσο όταν ξεκίνησε τη διαδρομή αυτής τη έκθεση πριν από λίγους μήνε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ Η κυρία Επίτροπος έχει το λόγο. Πρόεδρε, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω. Γιατί πραγματικά οι προεμπορικές δημόσιες συμβάσεις έχουν διπλό στόχο. Βελτιώνουν την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών και ανοίγουν τις ευκαιρίες για την ε, βιομηχανία να αναλάβει την ηγεσία στις διεθνείς αγορές. Είναι λοιπόν πραγματικά πολύ καλά δαπανημένα τα χρήματα αυτά και ένα παραπάνω σε, σε περίοδους κρίσης όπου θέλουμε η βιομηχανία μας να μπορεί να εφαρμόσει τα αποτελέσματα της έρευνας και να χρησιμοποιήσει κατά δυνατό καλύτερο τρόπο τις τεχνολογικές λύσεις και τις καινοτομίες. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ο εισηγητής κ. Σάρμπορ μας όπως και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή υποστηρίξει αυτό που έχουμε προωθήσει εδώ και αρκετό καιρό. Αλλά άλλο να βρίσκεται στον αγωγό και άλλο να βγει στο φως της ημέρας από τον αγωγό αυτό για να εφαρμοστεί στην πράξη. Και ελπίζω η έκθεση του Κοινοβουλίου να ε, αποδειχθεί το κίνητρο, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την πολιτική έρευνας και καινοτομίας. Ιδίως έτσι θα μπορέσουν να ζητηθούν πιο καινοτομικά προϊόντα στην Ευρώπη, πράγμα που θα αποτελέσει πάρα πολύ σημαντική διαφορά, όχι μόνο για τις ΜΜΕ και γι' αυτό χαιρετίζω την πρωτοβουλία αυτή και συγχαίρω για άλλη μια φορά τον κύριο Χάρμπορ για ε, την εργασία του. Ποια είναι τα συγκεκριμένα επόμενα βήματα που πρέπει να αναλάβουμε σαν μια άμεση απάντηση στις συγκεκριμένες συστάσεις της έκθεσης. Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η Κομισιόν στηρίζει δράσεις για να προωθήσει την ε, ε, διάδοση των ε, εμπειριών και να μπορέσουν να εφαρμοστούν αυτά τα προεμπορικά σχέδια ευρέω σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε ζητήσει στο πρόγραμμα, ε, στο πρόγραμμα έρευνας ε, υπαριθμών 7 και σε άλλα προγράμματα για να ενισχύσουμε αυτές τις εξελίξεις. Μέσω και μακροπρόθεσμα νομίζω ότι θα πρέπει στο μέλλον οι, ε, οι βουλές στην Ευρώπη να ενσωματώσουν τα στοιχεία αυτά στις δικές τους αγορές και θα πρέπει έτσι να ξεκινήσουμε εμείς από πλευράς Κομισιόν και θα ήθελα να το τονίσω σε μια εκείνες που βλέπετε για τον Μάρτιο τρέχοντος έτος που θα προτείνω μια ενδυναμωμένη στρατηγική για την ε, πληροφορική έρευνα και την ανάπτυξη στην Ευρώπη και μέσα στα πλαίσια των προεμπορικών δημοσίων συμβάσεων. Ξέρετε, ορισμένα κράτη-μέλη έχουν ξεκινήσει πειράματα με κάποια σχέδια για προεμπορικές ε, συμβάσεις αυτού του τύπου και θα ήθελα να καλέσω τα μέλη της Αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και όλου του σώματος να πάνε στις πατρίδες τους, να μιλήσουν στους υπουργούς, να μιλήσουν και στις ε, τοπικές αυτοδιοίκησεις όσον αφορά τις προεμπορικές ε, δημόσιες συμβάσεις και έτσι θα μπορέσουμε πραγματικά να πετύχουμε πολλά και ευχαριστώ που μας βοηθήσατε. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε και τον τελευταίο παρόντα βουλευτή απόψε για ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Η θα γίνει αύριο. Η επόμενη συνεδρία θα γίνει αύριο, Τρίτη, σε 9 το πρωί, το απόγευμα και το βράδυ. Η μεσαία διάταξη έχει δημοσιευθεί στον ανάλογο εγγράφο και στο ίντρανετ. Σας εύχομαι καλό βράδυ. Καληνύχτα.